Σας ευχαριστώ. Λοιπόν, αυτές ήταν οι ανακοινώσεις. Τώρα, οι αρμόδιες αρχές της Σουηδίας μου ανακοίνωσαν την αναπλούση της κυρίας Λένα Εκ από τον κύριο Κεν Τζόχασον ε, από την 18 Οκτωβρίου 2011. Καλωσορίζω τον ε, νέο συνάδελφο. Σας καλωσορίζουμε αγαπητέ συνάδελφε. Τώρα, σύμφωνα με το άρθρο 3 παράγραφος 2 του κανονισμού, μέχρι ότου δεν ελεγχθούν ε, τα, ε, ε, η ενεχθή εντολή, ο κύριος Τζόχασον είναι μέλος του Κοινοβουλίου με πλήρη δικαιώματα, με την προϋπόθεση φυσικά να έχει κάνει τη δήλωση ότι δεν ασκεί κάποια καθήκοντα ασύμβαστα με το έργο του Ευρωβουλευτή το διορθωτικό ε, σύμφωνα με το άρθρο 216 του κανονισμού η Επιτροπή Μεταφορών